Και εδώ λίγη η συζήτηση και προχωρούμε στις αγορεύσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 60, 163 του κανονισμού. Και πρώτη κυρία Ισταράς Φεραγκούτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει το θέμα της ευρωπαϊκής ρύθμισης για την προσβασιμότητα και συστήνει στα κράτη-μέλη κάποια ελάχιστα επίπεδα έτσι ώστε τα, οι πολίτες ε, με προβλήματα κινητικότητας ε, να μπορούν να μετακινούνται χωρίς εμπόδια στις μεταφορές, στις νέες τεχνολογίες και τα λοιπά στον τόπο εργασίας τους, στην κατοικία τους και θα πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις της κοινωνικο-οικονομικές τις οποίες θα έχουν τα μέτρα αυτά για τα πρόσωπα που έχουν τέτοια προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο ε, θα ε, τεθούν σε λειτουργία τα μέτρα αυτά. Ε, δεν έχουμε, έχει υπάρξει μια μελέτη από το 2012, αλλά δεν γνωρίζουμε τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής και θα πρέπει να μας διαθέσει τη μελέτη έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταθμίσουμε ε, τις εξελίξεις, ε, τις θετικές, ε, για να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρίες. Ευχαριστώ κυρία Εστάρας Φεραγκούτ. Ο κύριος Γέρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνω έκκληση στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Τούσκ. να μην κλείσει τα πολωνικά ανθρακοριχεία που αποδίδουν φθηνή ενέργεια. Πρέπει να το κατανοήσει αυτό η πολωνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υποχωρήσει απέναντι στις πιέσεις των λόμπι. Πρέπει να προχωρήσει μια πραγματική ενεργειακή ένωση που μπορεί να βασίζεται και στον άνθρακα, αλλά βέβαια και σε κοινέ διαπραγματεύσεις για τις τιμές του φυσικού αερίου. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεκ. Ο κύριος Λούκε. Μπεν Λούκε. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα προχώρησε εκλογές και ο λαός μίλησε. Επί χρόνια φτιάξαμε ένα σύστημα κατεύθυνσης της οικονομίας με πολλά νομοθετήματα, συμφωνίες και συμβάσεις. Έρχεται ο ελληνικός λαός και λέει όχι, δεν δέχεται τα μέτρα που έρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκφράζει τη δική του θέληση. Αυτό σημαίνει όμως ένα πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το χειρίζεται αυτό εν του γεγονότος ότι εδώ εκφράστηκε δημοκρατικά η βούληση του ελληνικού λαού. Πώς είναι δυνατόν να επιμείνει το ευρωπαϊκό επίπεδο στην τήρηση των συμφωνημένων όταν ο ελληνικός λαός με δημοκρατικές εκλογές λέει «δεν θέλω». Δείχνει το πρόβλημα αυτό πόσο έντονη είναι η σύγκρουση μεταξύ των αξιώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάει να αναμειχθεί στα εσωτερικά των χωρών μελών και της βούλησης των λαών πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή της ευθύνης για τις ίδιες ενέργειες, για τις, την ανάλυση της ευθύνης για την ίδια οικονομική διαχείριση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Βίλαντ, ευχαριστώ κύριε Λούκε. Ακολουθεί τώρα ο κύριος Γιάκοφτσίτς. Σας ευχαριστώ. Αντίθετα με τον ε, Σλοβαίνο ε, Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος μιλάει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την ε, χρήση της, του όρου Τεράν για το κρασί της Κροατίας, εγώ θα ήθελα να έχουμε καλές γειτονικές σχέσεις και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα με πολιτισμένο τρόπο. Το Τεράν είναι ένα είδος ίνου, το οποίο καλλιεργείται στην ε, περιοχή εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Και παράγεται λοιπόν πολύ καλής ποιότητας ε, κρασί τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν όλοι και οι Σλοβενοί και οι Ιταλοί και οι Κροάτες που παράγουν το κρασί αυτό να κάτσουν να βρουν μια λύση. Εμείς από την Ίστρια λοιπόν δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη του κρασιού αυτού για μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιακόφτσης. Ο κύριος Φλάνακαν δεν είναι εδώ, γι' αυτό το λόγο έχει η κυρία Αλμπιόν Γκούσμαν. Εμείς τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αύξηση της καταστολής ε, και προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την κοινωνική διαμαρτυρία και γι' αυτό η κυβέρνηση και η οικονομική εξουσία αντιδρά με πάρα πολύ αυταρχικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν καταδίκες συνδικαλιστές ε, τέσσερα χρόνια καταδίκης, φυλάκισης, ε, πάρα πολλοί άλλοι έχουν επίσης καταδικαστεί σε, σε ποινές φυλάκισης ε, λόγω της ε, διαμαρτυρίες τους. Είναι 300 οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι υπόδικοι, συνδικαλιστές και διαμαρτυρόμενοι και η ισπανική κυβέρνηση δεν ε, παρέχει ε, θα έλεγα το δικαίωμα σε μια σωστή δίκη. Υπάρχει μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας και βίαιη μεταχείριση των κρατουμένων. Ευχαριστώ και εσάς, κυρία συνάδελφε. Κύριος Σκέρλεκ. Ευχαριστώ. Μιλώ εξ ονόματος των Κροατών πολιτών που ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο η κροατική κυβέρνηση ξεκίνησε και προχωρεί με τη διαδικασία Έρευνα για πετρέλαιο στις αδριατικές ακτές, στις Αδριατική. Τίθεται το ερώτημα του περιβάλλοντος και βέβαια και της παραγωγής τροφίμων που πάει και για τον κουρατικό λαό και για ευρωπαίους καταναλωτές. Ο οργανισμός πετρελαίου στην Κροατία δεν σέβεται τις αρχές που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν προχωρεί σε διαβουλεύσεις με άλλες χώρες της Αδριατικής Υποπεριφέρειας, αγνοώντας τα συμφέροντα των Κροατών πολιτών, αλλά εμποδίζοντας και άλλες κυβερνήσεις να σεβαστούν τα δικαιώματα των πολιτών τους. Ζητώ λοιπόν να του υπομνηστεί, να υπομνηστεί στην κρατική κυβέρνηση η ανάγκη να σέβεται τις αρχές αυτές. Ευχαριστώ. Τώρα ακολουθεί ο κύριος Κοράου. Θα ήθελα να πω ότι εμείς εμένουμε να θεωρούμε την δραστηριότητα της μαφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κάτι το μη σημαντικό. Αυτό το φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε με ευκαιριακό τρόπο σε διάφορες επιτροπές πρέπει να γίνει η απόλυτη προτεραιότητα γιατί τροφοδοτεί τη διαφθορά, τροφοδοτεί την τρομοκρατία και δημιουργεί καταστάσεις απαράδεκτες, δυστυχέστατες, οι οποίες ε, ε, προκαλούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τη δράση μας και μέσω μιας ειδική εισαγγελία για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Θα μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε και ένα μέσο το οποίο μπορεί ε, να διασφαλίσει την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και να κόψει την τροφοδοσία αυτών των οργανώσεων που είναι η φτώχεια. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Κοράου. Ο κύριος Παπαδάκης. Τα μέτρα της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης Draghi και του επενδυτικού πακέτου Juncker προσφέρουν κρατικό χρήμα στα μονοπόλια και καταδικάζουν στη φτώχεια τους λαούς την ίδια γραμμή στηρίζει η νέα κυβέρνηση σύριζα ανεξάρτητοι Έλληνε στην ελλάδα διαβεβαιώνοντας ότι θα τηρήσει τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και του νατο και θα προωθήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση ονομάζοντας κοινικά τη φτώχεια του λαού λιτό βίο. γι' αυτό λοιπόν δεν συνιστά αλλαγή υπέρ του λαού η κυβερνητική αλλαγή στην ελλάδα το κκε και με την ενίσχυσή του στι εκλογές θα προσφέρει όλες του τι δυνάμει ώστε ο λαός να μην δείξει ανοχή στην κυβέρνηση και να σηκώσει ανάστημα για την ανάκτηση των απολειών του με μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση να αναμετρηθεί με τον πραγματικό αντίπαλο την ευρωπαϊκή ένωση τα μονοπόλια και την εξουσία του. Σα ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Παπαδάκη. Ο κύριος Στικόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, για πολλούς ε, ανθρώπους η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου θέλουν να ζήσουν όλοι. Το δίχως άλλο. Για μένα οι σκανδιναβικές χώρες είναι ενδιαφέρουσες. Ε, αλλά διαπιστώνουμε ότι στην Νορβηγία ετησίως εκατοντάδες παιδιά πολύ απλά τα παίρνουν από τους γονείς τους. Πόσο θα κλείνουμε λοιπόν τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Εγώ ίδιος διαπίστωσα ότι δεν φτάνει για την περίπτωση αυτή να χρησιμοποιηθούν μόνο νομοθετικά μέτρα και τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα. Υπάρχει η Εύα Μιχαλάκοβα, για παράδειγμα, μια γυναίκα από την Τσεχική Δημοκρατία την οποία και κατηγορούν χωρίς να έχει αποδεχτούν, να έχουν αποδεχθεί αυτές οι κατηγορίες και πολύ απλά τις αφορούν τα παιδιά της, τις θα τα παιδιά της. Ερωτώ λοιπόν πόσο θα αγνοούμε αυτό το φαινόμενο με τους Τσέχους πολίτες ε, για την Νορβηγία και τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Σάιμον. Micro. Η εκλογική μου περιφέρεια των West Midlands βρίσκει να της λείπουν 718.000 λίρες από ευρωπαϊκά χρήματα λόγω της αναζωνίας και μυσαλλοδοξίας της Βρετανικής συντηρητικής κυβέρνησης. Όλες οι άλλες χώρες μέλη, όλες οι περιφέρειες έχουν συμφωνήσει το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο η συντηρητική κυβέρνηση δεν θέλει να συμφωνήσει. Στα West Midlands μιλούμε για 140 εκατομμύρια για την Black Country 201 εκατομμύρια λίρες για την ευρύτερη περιοχή του Μπίρμιχα, 170 εκατομμύρια λίρες για άλλες περιοχές της εκλογικής μου περιφέρειας, τα οποία δεν λαμβάνουμε και την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση των Τόριδων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη Γερμανία. Το οποίο ενδεχομένω να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για εσά, κύριε Πρόεδρε, γιατί από 1η Ιανουαρίου του τρέχοντο έτου υπάρχει ε, ένα νόμο στη Γερμανία για του ελάχιστου μισθού, για του κατώτατου μισθού, που θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτόν και οι μεταφορικέ εταιρείε. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό ο νόμο, τουλάχιστον 1,8 ευρώ ανά ώρα. Αυτό είναι τετραπλάσιο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά στην Τσεχία και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στην κατάσταση αυτή ότι αυτό το κατάστατος μισθό είναι αντίθετο με την εσωτερική αγορά. Γιατί έτσι δημιουργείται εμέσως εμπόδιο στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κάτι να κάνει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι καθόλου σαφές κατά πόσον αυτό επιτρέπεται καν νομικά να ισχύει αυτό και για τις εταιρείε μεταφορών. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Ζαχραντήλ. Και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Πάετ. Δεν ξέρω αν σωστά το προφέρω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα χωρίς να αναφερθώ στην κατάσταση στην Ουκρανία, γιατί η σύγκρουση στην Ουκρανία θα πρέπει κατεπηγόντως να ε, έχει διεθνή παρέμβαση για να απαιτευθεί νέα και χειρία και να επιτρέψει μια ερνηστική δύναμη στην χώρα. Αυτό το βήμα θα τερμάτιζε τη βία και την απώλεια περαιτέρω επικράτεια της Ουκρανίας. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι στους πρόσφατους μήνες ε, είχαμε διάφορες καταστάσεις ε, με αεροπλάνα πολιτικά και στρατιωτικά τα οποία πετούν χωρίς πομπολίπτες και ιδιαίτερα στην ε, περιοχή της Βαλτικής. Και αυτό σημαίνει ότι όταν ε, ταξιδεύουν με κλεισμένα τα συστήματα επικοινωνίας τους, τα αεροπλάνα αυτά αποτελούν κίνδυνο για τους επιβάτες τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει η σχετική νομοθεσία για τα σχετικά αεροπλάνα προκειμένου να επιβάλλεται η χρήση τέτοιων πομπολιπτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο να μιλεί κανεί για πόλεμο και για τις φρικιαστικές του συνέπειες και βέβαια και δαπανηρή υπόθεση. Εγώ είχα την ατυχία να υποχρεωθώ να υπηρετήσω το ρωσικό στρατό στη δεκαετία του 80. Είναι δαπανηρή η ουκρανική κρίση. Έχει μειωθεί το ε, εθνικό εισόδημα, έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το ερώτημα είναι τελικά έχουμε αναλάβει τις απαραίτητες δεσμεύσεις για διάφορα είδη βοήθειας προς την Ουκρανία. Θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες κρίσεις γύρω-γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η Παλαιστινιακή Αρχή λαμβάνει 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και τώρα υπάρχει και πρόταση της Γερμανίδας Καγκελαρίου να διαθέσει το ίδιο ποσό στην Ουκρανία. Όμως εκεί το μέγεθος της οικονομίας της χώρας αυτής είναι πολύ διαφορετικό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Τάραντ, ακολουθεί ο κύριος Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Τουρκία εδώ και 40 χρόνια κατέχει χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχει ουσιαστικά ευρωπαϊκό έδαφο, δημιουργώντα τραγικέ συνέπειε, οι οποίε συνέπειες καταγράφονται ω 200.000 πρόσφυγε Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτε, οι μοναδικοί Ευρωπαίοι πολίτε πρόσφυγε, αλλά υπάρχουν ακόμα και πιο τραγικέ πτυχέ αυτή τη τραγωδία, όπω είναι οι αγνοούμενοι. Δυστυχώ η Τουρκία και γι' αυτό το εξαιρετικά ανθρωπιστικό θέμα αντί να επιδείξει ευαισθησία επιδεικνύει το ίδιο απάνθρωπο πρόσωπό τη. αρνείται πεισματικά να ανοίξει τα αρχεία του τουρκικού στρατού για να μπορέσει να εξευρεθεί η τύχη αυτών των αγνωμένων. ταυτόχρονα ορισμένε στρατιωτικέ περιοχέ τι χαρακτήρισε ούτω καλούμενε στρατιωτικέ περιοχέ για να απαγορεύει την ανέβρεση των αγνωμένων. ταυτόχρονα έδωσε, εκτέλεσαν ψυχρό το 1974 70 άμαχου από την κοινότητα Νάσσα, του οποίου μετέφεραν κάπου αλλού και δεν καταμαρτυρούν σήμερα που βρίσκονται. Εμεί καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα απέναντι σε αυτήν τη χώρα υποένταξη για μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω είναι η Κύπρο. Επιτέλου η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει για αυτό το. Ευχαριστώ κύριε Χριστοφόρου. Η Το στρατηγικό αυτό πρόγραμμα επενδύσεων πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπως το έχει ήδη πει ο πρόεδρος Γιούνκερ. Γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε απευθείας τους πολίτες, θα πρέπει να βρούνε τον τρόπο οι πολίτες για να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους, να νιώσουν ότι τους ανήκει η ευρωπαϊκή διαδικασία, να βρούμε νέες μορφές χρηματοδότησης του Ταμείου, μικροδωρεές, το λεγόμενο crowdfunding του διαδικτύου, έτσι ώστε οι πολίτες ε, να επηρεάσουν ε, <clears throat> την ίδια τους τη ζωή όπως το έχει κάνει σαν παράδειγμα το πρόγραμμα Εράσμος. Έχω λάβει πάρα πολύ ενθουσιώδεις απαντήσεις από τους νέους γι' αυτό. Υπάρχει μια επιθυμία για την Ευρώπη ε, στους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά δεν έχουμε τους σωστούς τρόπους για να διοχετεύσουμε την επιθυμία αυτή. Απαιτείται θάρρος και τόλμη. Ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε σοβαρή παραβίαση πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας, των πολιτών του Γιβραλτάρ. Υπάρχει η πρόταση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, που περιλαμβάνονται διατυπώσεις για το γεγονό ότι η πρόταση θα εφαρμόζεται πλήρως και στο Γιβραλτάρ. Όμως πέρασε μετά το 2014 πρόταση για τον αποκλεισμό του Γιβραλτάρ και των πολιτών του. Αυτό είναι απαράδεκτο. Φανταστείτε να είχαμε αποκλείσει κάποιους Ευρωπαίους πολίτες στην βάση του φίλου τους ή της εθνικότητάς τους. Και όμως το κάνουμε αυτό τώρα στη βάση εθνικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν μπορεί πλέον να υποφελείται από την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ελευθερία των Ουρανών μετά από ένσταση της, Ευρω... της Ορίστε που έχουμε φτάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο πρόεδρος Βίλαντ, ο κύριος Βάιγκελ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Πράγματι σε ένα τμήμα πολύ ευαίσθητο της Ευρώπης εξακολουθεί να μένεται ένας πόλεμος. Ενθυμίστε εδώ και χρόνια που βλέπαμε στα νέα στις ειδήσει ε, τους, τις μάχες στα Βαλκάνια. Δυστυχώς όμως οι εικόνες αυτές επανέρχονται. Πάρα πολλοί ε, αναζητούν να βρουν λύσεις για να ξεφύγουν από τους πολέμους και αυτή είναι φυσικά η άμαχη των συγκρούσεων αυτών. Θα υπάρξει λοιπόν μια νέα γενιά παιδιών προσφύγων. Δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε αυτό με τις διαπραγματεύσεις ή με άλλο τρόπο, με άλλα μέτρα, εν πάση περιπτώσει μέτρα πιο αποτελεσματικά για την προστασία των αμάχων. Ο πόλεμος ε, δεν κάνει διακρίσεις, ε, τα θύματα πολλές φορές είναι εντελώς αθώα. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει κ. Καλινόφσκι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 19 Ιανουαρίου το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας μας ενημέρωσε για διμερή συμφωνία την οποία και συνήψε με την Ρωσική Ομοσπονδία για την εξαγωγή χοιρινού. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των, ανθρωπίν, των ευρωπαϊκών κανόνων. Το ήξερε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει τη διαδικασία αυτή η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία είναι θέμα ύψης της σημασίας. Αν η Ρωσική Ομοσπονδία έχει δοκιμάσει πολλές φορές να διασπάσει την ενότητά μας, εμείς έχουμε επιβάλει το εμπάργκο στην εξαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων προς τη Ρωσία και έχουμε ε, εμπλακεί στην ε, σύγκρουση στην Ουκρανία. Ξέρουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι το ίδιο στοιχείο, το ίδιο θέμα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να διασπαστεί η ομόνια μας και καλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το φροντίσει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε Καλινόφς, τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος Κρυμπαν Ντάλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Το 1984 ε, κάποιοι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Camel Lerd ε, καταδικάστηκαν λόγω της δράσης τους και δεν αθώθησαν από τότε. Ένας από αυτούς εξήγησε πέρυσι ότι παρά το ότι ε, δεν παραβίασαν κανένα νόμο, παρόλα αυτά δικάστηκαν οι απεργοί των ναυπηγείων Camel Lerd, είχαν υπάρξει και άλλες κακοδικίες αν θέλετε ε, στη χώρα μου που είχαν επιβληθεί από τους υπουργούς εκείνης της εποχής για να ε, αυξήσουν τα επίπεδα καταστολής. Η πρόσβαση στα επίσημα αρχεία είναι απαραίτητη για αυτούς οι οποίοι ζητούν τη δικαίωσή τους. Είχαν παραβιαστεί τα δικαιώματα των εργατών του ναυπηγείου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πιέσει έτσι ώστε να αποδεσμευτούν τα έγγραφα και να δικαιωθούν επιτέλους οι εργαζόμενοι σε αυτήν την επιχείρηση. Ευχαριστώ κύριε Ντάβλιν. Μάτω. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν θα μιλήσω για το ισπανικό Ιμπλατάρ, θα μιλήσω όμως ε, για τις επενδύσεις στην έρευνα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε τον καλύτερο αστρονομικό ουρανό της Ευρώπης, ιδιαίτερα στις Κανάριες νήσους. Εδώ και 30 χρόνια συνεργάζεται με πάρα πολλά ερευνητικά ιδρύματα, κυρίως της Ευρώπης απαιτείται περισσότερη συνεργασία έτσι ώστε ε, να πάρει μέρος στο νέο πρόγραμμα του μεγάλου ε, τηλεσκοπίου ε, με ακτίνες γάμα, το μεγαλύτερο του πλανήτη πρέπει να ενισχυθεί και από την Ισπανική κυβέρνηση, κάτι το οποίο θα βελτιώσει τις δυνατότητες της επιστήμης και της έρευνας στην Ευρώπη. Το νέο αυτό τηλεσκόπιο θα είναι ένα ποιοτικό άλμα για την επιστήμη. Ε, ζητώ λοιπόν την στήριξη του προγράμματος του αστροφυσικού αυτού παρατηρητηρίου. Σας ευχαριστώ αδελφέ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ροντρίγκες Φερνάντες. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επένδυσε ε, πάρα πολλά στην περιοχή της Βαλένσια για την ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Κάποια χρόνια μετά βλέπουμε ότι έχουν καθυστερήσει οι μεταρρυθμίσεις, κάποια σχολεία δεν έχουν πάρει ακόμα τίποτα και πάρα πολλοί ε, μαθητές σπουδάζουν κάτω από απαράδεκτες κτηριακές συνθήκες εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε από τη δική της πλευρά η τοπική αρχή της Βαλένθια να φέρει εις πέρας και να σεβαστεί τις ανηλυμένες της υποχρεώσεις. Γιατί υπάρχουν μαθητές οι οποίοι για 8 χρόνια σπουδάζουν σε καλύβες θα έλεγε κανείς και σε πρόχειρα καταλήματα. Η τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια δεν ήταν σε θέση ε, να φέρει πέρα στις υποχρεω... να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, ε, έκανε απολύσεις μόνο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν με αρνητικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Επόμενος είναι τώρα ο συνάδελφος Βαλάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης του Συμβουλίου των Υπουργών ε, Γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν επιτρέπεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την πώληση γυρνού κρέατος. Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Η Ρωσία θέλει να προκαλέσει κατακαιρματισμό της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να επιτρέψουμε διακριτική μεταχείριση κατά οποιοδήποτε κάτω μέλους. Σε ό,τι αφορά τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά και σε περιπτώσεις κρίσης, ιδιαίτερος εν ώψη της κατάστασης στην Ουκρανία, θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και ομόνια. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Βαλέσσα, και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Νέκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις στον κόσμο που οδήγησαν στη μετακίνηση 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. τα τελευταία δύο χρόνια 18 εκατομμύρια μετανάστες αναζήτησαν καταφύγιο στη Βουλγαρία και δεν λειτουργεί σωστά το Δουβλίνο 2. Η κατάσταση για τη χώρα μου είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί όλοι αυτοί στην ουσία παραμένουν στο έδαφος της πρώτης χώρας μέλους στην οποία μπόρεσαν να φτάσουν. Τίθενται λοιπόν κάποια θέματα σημαντικά για τη χώρα μου, όπως η ολοκλήρωση του χώρου Σέγγεν της, ε, με τη Βουλγαρία, και τα δικαιώματα των προσφύγων. Αυτά συνδέονται με το θέμα του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της χώρας και θα πρέπει να τύχουν εξέτασης από την ε, Επιτροπή. Η είσοδος της Βουλγαρίας στο χώρο Σέγγεν είναι προτεραιότητα, όχι μόνο για την ίδια τη Βουλγαρία, αλλά και για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Νεκόφ. Κύριε Σόιντροβα. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας συμβαίνει κάτι το ανησυχητικό. Η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε έγγραφο όπου κατηγορεί έναν Πρίτανη της σχολής για προπαγάνδα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα γνωρίζουμε από τις εποχές του απολυταρχισμού, ότι έκανε προσπάθεια δηλαδή να ελέγξει τις ανώτατες σχολές. Και μάλιστα οι κατηγορίες αυτές απευθύνθηκαν στον ε, Πρίτανη αυτόν και ενώπιον των φοιτητών Ζητώ να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει εντολή στις αντιπροσωπείες της στην Ρωσία, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Ο κύριος Μπρέναν. Την προηγούμενη Παρασκευή πήγα σε γαλακτοπαραγωγούς στην εκλογική μου περιφέρεια στην Βόρειο-Ανατολική Αγγλία και συναντήθηκα εκεί με γαλακτοπαραγωγούς, τον Ρίτσαρτ και τον Ντένις που έχουν 300 αγελάδες στο αγροκτημά τους και ως αποτέλεσμα της πτώσης του, της τιμής του γάλακτος τους τελευταίους μήνες ε, σημειώνουν τώρα σημαντική πτώση στο εισόδημά τους. Αυτό πλήττει όλους τους γαλακτοπαραγωγούς στο Ενωμένο Βασίλειο. Και τι πρέπει να γίνει τώρα Κάτι που μπορούν να κάνουν οι πελάτες είναι να ζητήσουν από τη διεύθυνση των σούπερ μάρκετ όπου πηγαίνουν να ψωνίσουν να μάθουν αν πληρώνουν έντιμες τιμές στους παραγωγούς. Πίεση των καταναλωτών. Σωστά κάνουν και αρμέγουν τις αγελάδες τους γαλακτοπαραγωγή, αλλά όχι να αρμέγουν τα σούπερ μάρκετ, τους γαλακτοπαραγωγούς και τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρέναν. Τελείωσαν εδώ οι αγορεύσεις του ενός λεπτού. Έχω δύο ανακοινώσεις από την ομάδα των συντηρητικών. Έλαβα την ε, ειδοποίηση ότι αντικαθιστά ο κύριος Μπασίρ, τον κύριο Καμάλ, ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Δεύτερη ανακοίνωση που έχω είναι ότι ο κύριος Γιώργος